Καλό σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε, μάλλον να επανέλθουμε, σχετικά με την εκρίζωση των στερεοτύπων για τα φύλλα, σχετικά με την ταυτότητα του να είσαι αρσενικός. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζω σε αυτό το εργαστήριο για τα πολιτικά δικαιώματα και τα θεσμικά ζητήματα για την Επιτροπή Γυναικών. Ξεκινάμε με μια ανακοίνωση πρακτικού περιεχομένου. Πρέπει να σας πω ότι η κυρία Κέιτ Ντόιλι αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή της για ιατρικούς λόγους, για λόγους υγείας, και λόγω της ανακοίνωσης αυτής που έγινε τελευταία στιγμή δεν μπορέσαμε να την αντικαταστήσουμε. Έχουμε όμως τρεις διακεκριμένους εμπειρογνώμονες μαζί μας σήμερα και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ε, παρεμβάσεις τους. Την τελευταία δεκαετία ο ρόλος των ανδρών έχει προκύψει ως σημαντικό ζήματα στα θέμα, ζήτημα με στα θέματα ισότητας των φύλων πολύ συχνά με τα θέματα ισότητας των φύλων ως ζήτημα των γυναικών καθότι ήταν αυτές η κινητήριος δύναμη πίσω από την όθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων και γενικώ στην κοινωνία. Από την άλλη μεριά έχει, δίνεται όλο και μεγαλύτερη σημασία στην κατανόηση των ανδρών του ζητήματος της ισότητας των φύλων η ταυτότητα αυτή της αρενοπότητος σε βάση περιπτώσει συμπεριλαμβάνεται όλο και πιο συχνά σε σχετικές μελέτες για μια πιο ισότιμη δίκαιη κοινωνία. Αλλά έχουμε περιορισμένη συστηματική γνώση σχετικά με το θέμα αυτό στις διάφορες χώρες μέλη. Στο εργαστήριο αυτό θα επιχειρήσουμε να καλύψουμε κάποια από τα κενά αυτά και να παράσχουμε τροφή προς σκέψη. Η κυρία Κάμπορα, να ακούσαμε καλά το όνομά της, είναι από το κέντρο μελετών του Γκράτσα της Αυστρίας για τον ρόλο των ανδρών στα θέματα ισότητας των φύλων. Και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. στο εργαστήριο αυτό για την εκρίζωση των στερεοτύπων σχετικά με το ρόλο των ανδρών στα θέματα ισότητας των φύλων. Με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα της μελέτης που είχαμε για τα θέματα ισότητας των φύλων και στα οποία συμμετείχα. Θα εστιαστώ στο θέμα της φροντίδας σχετικά με την αρινοπότητα Όπως και στο ρόλο των γυναικών στην οικονομική μεγέθυνση που μπορούμε να έχουμε με καλύτερη απορρόφηση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σταδιακά, ο ρόλος των ανδρών και το ζήτημα της ισότητας των φίλων... τίθεται όλο και πιο επιτακτικά, με όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση ότι η συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα, την οικογενειακή και ο ρόλος των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα αυτό και με μελέτες που είχαμε ζητήσει σχετικά με την ισότητα των φίλων εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το ρόλο των φίλων με κάποια δεδομένα που προκύπτουν από τις μελέτες αυτές για τους άνδρες. Δουλεύει αυτό, λέει η ομιλήτρια. Έδειξε λοιπόν η μελέτη ότι οι άνδρες όλο και περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και δεν μπορεί πλέον να θεωρείται περιθωριακός ο ρόλος τους στη φροντίδα των παιδιών. Αν και ακόμα και οι πιο προχωρημένες κοινωνικά χώρες στην Ευρώπη απέχουν από μια χρηστή ισορροπία. Αυτό ήταν μια από τις βασικές από τα βασικά πορίσματα της μελέτης. Οι όποιες λύσεις μπορούν να δοθούν εξαρτώνται από τα θέματα αντίληψης της ότως των φύλων, από τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και της αντίληψης του ρόλου τους, όπως και από διατάξεις κοινωνικής πρόνοιας. Και καθότι, μάλλον παρότι οι άνδρες αυξάνουν το μερίδιο της συμμετοχής φροντίδας στο σπίτι, πρέπει να εξετάσουμε ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις της τάσεως αυτής και ποια εμπόδια υπάρχουν. Ας μιλήσουμε πρώτα για το γενικότερο πλαίσιο. Όπως είπατε πρόεδρε, πολύ καιρό στο παρελθόν οι πολιτικές ισότητες των φίλων εστιάζονται στις γυναίκες. Λάβαμε σημαντικά βήματα προκειμένου να ξεπεράσουμε ένα διανοητικό μπλοκάζ που είχε εμφανιστεί σχετικά με την αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα αυτά. Το gender mainstreaming έχει βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων αυτών και στην καλύτερη κατανόηση και αντίληψη από πλευρά των ανδρών του ρόλου που διαρματίζουν στην οικογένεια. Με διάφορα συνέδρια και παρουσιάσεις που είχαμε στις σκανδιναβικές χώρες μεταξύ άλλων όπου ενθαρρύνθηκε ο ρόλος των ανδρών στη φροντίδα που παραέχουν και στο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν περαιτέρω. Επρόκειτο για την πρώτη συστηματική εξέταση όλων των κρατών μελών σχετικά με θέματα κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας και εκπροσώπησης. in the uh, last Τι άλλαξε λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες. Η όλο και αυξανόμενη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών η αλλαγή των προτύπων στην παροχή φροντίδας οικογενειακής μας οδηγούν στο να εξετάσουμε την πραγματική συνεισφορά των ανδρών στις περισσότερες από τις εβραϊκές κοινωνίες. Η φροντίδα παραμένει στις περισσότερες από τις εβραϊκές χώρες ένα ζήτημα βαθιά αγκυρωμένο στην αντίληψη του φίλου, αλλά και στην αντίληψη της κοινωνικής τάξης, της εθνικότητος κτλ οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο αν αντιληφθούμε και αναγνωρίσουμε την αλλαγή του ανδρικού ρόλου στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας που ήταν εμπόδιο στο παρελθόν για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών έχουν υπογραμμιστεί. Και εδώ μιλούμε κυρίως για την φροντίδα των παιδιών. Υπό την έννοια της ισότητας των φύλων, δεν θα ήταν επιθυμητό η φροντίδα αυτή να παραμείνει ζήτημα των γυναικών. Και υπό την έννοια των δημογραφικών αλλαγών που παρατηρούμε, μάλλον δεν είναι πιθανό κάτι τέτοιο. Ας περάσουμε τώρα σε κάποια σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Οι μελέτες που έχουμε αναθέσει μας δείχνουν ότι η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μεταξύ των φύλων, μεταξύ του 2000 και του 2010, έχει πάει σε κάποια θέματα σύγκλησης σε σχέση με την αγορά εργασίας. Δηλαδή σε αυτή τη δεκαετία το κενό απασχόλησης μειώθηκε το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών με μια σχετική αύξηση της δεύτερης κατηγορίας και σχετική μείωση της πρώτης. Ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί και για τους δύο, και για τις δύο ομάδες, αλλά περισσότερο για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες. Και αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση στη μελέτη. Έχουμε λοιπόν μια αυξανόμενη σύγκληση των τάσεων απασχόλησης των δύο πληθυσμών λόγω μιας κρίσης που έπληξε τομείς που παραδοσιακά ελέγχοντο επικυριαρχούντο από τους άνδρες. Στη βιομηχανία, στις ζώνες της υπαίθρου με έντονες απώλειες θέσεις απασχόλησης. Η ανδρική ταυτότητα που ήταν απολύτως συνδεδεμένη με αυτόν που κέρδιζε τα χρήματα για τον οικοκυριό δεν μπορεί πλέον να υλοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο γιατί από την πλήρη επασχόληση και τα σχετικά μοντέλα έχουμε περάσει σε άλλα μοντέλα μερική επασχόλησης. Ευελιξία και ανασφάλειας εργασίας. Επομένως, οι προσδοκίες του ανδρικού πληθυσμού να εξασφαλίσει μόνιμη απασχόληση έχει πληγεί. Και αυτό έχει πλήξει το μοντέλο του κυρίαρχου ρόλου αυτού που κερδίζει βασικά τα έσοδα της οικογένειας. Από τον πρωταρχικό ρόλο που είχαν οι άνδρες σε αυτό το πρότυπο, στο πρότυπο με μετακινήθηκαν σε ένα πρότυπο χαμηλότερων εσόδων και μεγαλύτερου μερίσματος εισφοράς φροντίδας ε, στις οικογενειακές ανάγκες το οποίο σχετίζεται και με διάφορες αντιλήψεις ηγεμονικού ανδρικού ρόλου εντός της οικογένειας. Έχουμε εμπειρικές ενδείξεις για την αλλαγή του ρόλου αυτού. Εδώ έχουμε ένα γράφημα. Έχουμε μια εμπειρική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης στον χώρο εργασίας και του χρόνου απασχόλησης στην εργασία. Αυτή το, αυτό το σχετισμό βλέπουμε στο γράφημα τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίηση είναι σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία με αντίστοιχα ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, ενώ η χαμηλότερη ικανοποίηση παρατηρείται σε χώρες με υψηλότατα όρια εβδομαδιαίας απασχόλησης. και εξαρτάται πώς προσμετρά κανείς τη μη πληρωμένη εισφορά των ανδρών σε εργασία, σε δουλειά, σε υπηρεσία φροντίδας. Εξακολουθεί να αυξάνεται αυτό σε κάποιες βόρειες χώρες και μειούται σε κάποιες πρώην σοσιαλιστικές, λέει ομιλήτρια, χώρες. Εξού και έχουμε το διπλάσιο σε κάποιες βόρειες χώρες από ό,τι σε κάποιες πρώην σοσιαλιστικές. Το θέμα είναι ποιος τελικά στην πραγματικότητα παρέχει τη φροντίδα. Ποιοι είναι οι άντρες εκείνοι που το πράττουν αυτό. Έχουμε λεπτομερείς έρευνες από το 2007 από την Ορβηγία, από, από το Ινστιτούτο Χόλτες Βάρεν Έγκελαντ, το οποίο βεβαίως προσμετρούσε ζευγάρια, ζεύγη, άνδρες υψηλότερου μορφωτικού επίπεδου είναι κατά ένα τρίτο πιο πιθανό να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο εισφοράς φροντίδας από τους αντίστοιχους χαμηλότερου μορφωτικού επίπεδου. Επίσης, άνδρες με υψηλότερα έσοδα μισθό είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο φροντίδας, ιδιαίτερα αν οι σύντροφοί τους έχουν χαμηλά έσοδα ή δεν έχουν απασχόληση. Και η πιο ισότιμη σχέση ήταν πιο έντονη και πιο εμφανής μεταξύ των νεαρών ζευγαριών παρά μεταξύ των ζευγαριών υψηλότερης ηλικίας. Ποιοι είναι οι λόγοι και οι αιτίες για τις διαφορετικές αυτές διαφορετήσεις. Κάποια ζευγάρια προτιμούν υψηλότερα επίπεδα εσόδων για τους άνδρες, ενώ άλλα ζευγάρια δίνουν προτεραιότητα στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα την οικογενειακή. Δηλαδή έχει αντικατασταθεί το πρότυπο εν μέρη αυτού που βασικά κερδίζει τα οικογενειακά έσοδα προς μια πιο ισορροπημένη κατάσταση, αλλά εξακολουθούν οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο εισφορά φροντίδα. Χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάποιες χώρες οι δεξιότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε μεγαλύτερη προσκόλληση στην παραδοσιακή αντίληψη της ε, δραστηριότητας των γυναικών στο σπίτι Δηλαδή έχουμε και κάποιες τάσεις σε κάποιες χώρες επανόδου στα παραδοσιακότερα πρότυπα του ρόλου των φίλων. Για κάποιους άνδρες το πράγμα είναι περισσότερο πρακτικό παρά θέμα νομοθεσίας ή κάποιου άλλου, κάποιες άλλες ε, ρήτρας που, τους, ε, που θα τους απαγόρευε ή θα τους καθοδηγούσε σε μια χαμηλότερη προσφορά φροντίδας. Επίσης το θέμα της άδειας πατρότητος δίνει κάποιες δυνατότητες, κάποιο περιθώριο στις οικογένειες. Γιατί ποικίλει πάρα πολύ στην Ευρώπη από μηδέν ημέρες μέχρι κάποιους μήνες αναγκαστικής άδειας όπως στην Ισλανδία, να ακούσαμε καλά την ομιλήτρια. Παρέχονται λοιπόν κάποιες ημέρες άδεια είτε πληρωμένες είτε μη πληρωμένες. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ διαφορετικό σύνολο εικόνα στις διάφορες χώρες. Οι άνδρες λοιπόν συμμετέχουν τόσο πιο εύκολα όσο υπάρχει η ανάγκη της φροντίδας, όσο αυτό υποστηρίζεται από την ομοθεσία και από τις συντρόφους τους και όσο δεν παρεμποδίζεται από την εταιρική τακτική και πρακτική. Δηλαδή, από τους εργοδότες τους. Οι μελέτες μας δείχνουν διάφορες τάσεις που θα ήθελα να αναφέρω πρωτού ολοκληρώσω. Έχουμε λοιπόν κάποιες μελέτες που μας δείχνουν ότι η αντίληψη των ανδρών σχετικά με την παροχή της φροντίδας είναι πιο θετική σε κάποιες χώρες που έχουν επιτύχει καλύτερο επίπεδο κοινωνικής ισότητας, ισότητας των φύλων, παρά σε χώρες που έχουν πετύχει χαμηλότερα επίπεδα. Και κατέρχεται η τάση αυτή όταν υπάρχει υψηλότερη πίεση και άγχος για τον κυρίαρχο ρόλο του αρχηγού της οικογένειας, αυτού που κερδίζει τα βασικά έσοδα που παρέχει για την οικογένεια. Κάποιες χώρες έχουν ενισχύσει την επιστροφή στο σκληρό μοντέλο της αρσενικής ταυτότητος και που σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει στις παροχές και ε, περιθώριο που παρέχουν στους πατέρες στην κοινωνία. έχουμε μια συγκριτική επίση μελέτη μεταξύ Νορβηγία και Πολωνίας που είναι ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει χαμηλότερε πιθανότητες ε, κρουσμάτων βία σε νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ισορροπία εσόδων. Εσόδων και ε, ε λήψης απόφαση σχετικά με τα οικογενειακά θέματα και την φροντίδα των παιδιών. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν δούμε την ισότιμη διαδικασία λήψεων αποφάσεων και τις πιθανότητες κρουσμάτων βίας, αυτά είναι και τα δύο αρκετά χαμηλά, λέει ο Μιλήτρια. Η ισότιμη πρόσβαση, εν πάση περιπτώσει, στην ευθύνη αυτή, έχει σχέση με την πρόσβαση και στις άδειε, τις πληρωμένες ημί και στην αντίληψη που έχουν τα δύο φύλλα για το ρόλο τους. Δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν περισσότεροι από τους άνδρες ώστε να παρέχουν πρωταρχικές φροντίδες όπως αυτές που παρέχουν καθημερινά γυναίκες λέει η ομιλήτρια. Αυτό επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι οι άνδρες δεν συμμετέχουν τόσο άμεσα με θέματα όπως η φροντίδα των υπερηλίκων, των παππούδων για παράδειγμα, το οποίο αποκαλούμε στα πλαίσια της μελέτης άτυπη παροχή φροντίδας, και στο γράφημα φαίνεται ότι μιλούμε για ε, ομάδες ηλικίας πολύ υψηλής. Η φροντίδα λοιπόν των παιδιών ίσως να είναι ένα πρώτο σημάδι, μια πρώτη ένδειξη περαιτέρω αλλαγής Γιατί οι άντρες δεν είναι απλώς πατέρες, λέει ο ομιλήτρια. Η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στην τροφή του παιδιού ή στο να το βάζεις για ύπνο σημαίνει και συναισθηματική υποστήριξη είναι μια βαθύτερη φροντίδα στην ανάγκη του παιδιού. Πέρα από άλλα ζητήματα που χρειάζεται το σπίτι όπως ο κύκλος των φίλων, οι παππούδες, οι υπερήλικες κτλ. Επομένως όλα αυτά σχετίζονται με μια κοινωνική πραγματικότητα ευρύτερη, λέγει η ομιλήτρια. Και κάποιες συστάσεις πρέπει να υπογραμμίσουμε σχετικά με τον ρόλο των ανδρών. Πρέπει να εστιαστούμε στο επιμορφωτικό ζήτημα, που είναι ζήτημα κλειδί. Πρέπει να καταλάβουμε περισσότερα για τον συσχετισμό της αρενοπότητος και της παροχής φροντίδας. Αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί σε θέματα πολιτικής, σε θέματα πολιτικής ισότητας των φίλων. Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο διάλογο επί των ζητημάτων αυτών. Χρειαζόμαστε μια κριτική σκέψη και τοποθέτηση απέναντι στα πρότυπα που επικρατούν. Ακόμα και για την εκπαίδευση των παιδιών από την πολύ μικρή τους ηλικία από το δημοτικό. και χρειαζόμαστε και μια διατομιακή φεμινιστική προσέγγιση, λέει ο Μιλητρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την παρουσίασή σας, ε, κυρία Σάμπορ. Ε, τώρα έχουμε μια ομάδα διαφόρων, μια ομάδα από την Εθνοσυνέλευση της Νιγηρίας και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτες μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, στις ερωτοαπαντήσεις, αν το επιθυμούν και αν έχουμε χρόνο. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Christian Βεσκέ, Stakeholder Relations Officer του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα μεταξύ των φίλων από το Βίλνιους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ και που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το θέμα. Α, αύριο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που αντιπροσωπεύω εδώ σήμερα ε, θα δημοσιεύσει τα νέα αποτελέσματα ε, του δίκτυου για το 2017 για την ισότητα των φύλων. Για αυτούς που δεν ξέρουν ε, τι είναι αυτός ο δείκτης, αυτός μετρά την πρόοδο στην ισότητα μεταξύ των φύλων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τον έχουμε προσδιορίσει αρκετές φορές ε, από το 2005. Αυτά τα αποτελέσματα που θα μας δείξουν τις ποσοτικοποιημένες πληροφορίες και θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ιδέα ε, για την ε, ζωή των ανδρών και των γυναικών ε, στην Ευρώπη. Αλλά προτού σας αναφέρω μερικά από αυτά τα αποτελέσματα, θα αρχίσω με ένα επιχείρημα που είναι σημαντικό όταν μιλάμε για τα στερεότυπα σχετικά με τα φύλλα και με την αρενοπότητα με τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είναι ποσοτικοποιημένα δείχνουν τις στάσεις των συμπεριφορών των ανδρών και γυναικών που ήδη αντανακλούν την συμμόρφωση προς αυτά τα στερεότυπα. Θα πρέπει βεβαίως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια ποικιλομορφία μέσα στις ομάδες και στην, στις προσμονές και στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ατομικό που είναι οι επιλογές ζωής για τους άντρες και τις γυναίκες. Αλλά δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την, τους άνδρες, τα φύλλα ε, και ε, τις, τα στερεότυπα. Ε, θα ήθελα να σας πω για κάτι ε, με το οποίο ασχολούμαι από τότε που ε, εξετάζω το θέμα σχετικά με το φύλλο. Έχουμε τον Herbert Meads που λέει ότι υπάρχει ένα συνέστημα καινού, ένα συνέστημα του μη ανήκειν, του ότι κάποιος δεν έχει θέση, έχει έλλειψη ταυτότητας, έλλειψη δομημένου όντως και εγώ. Έχουμε λοιπόν ένα άγχος που προκαλείται από αυτήν την κατάσταση και θα πρέπει να, το λάβουμε, να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη όταν μιλάμε για την αρενοπότητα. Τι είναι η αρενοπότητα? Είναι μια σειρά αντιφάσεων ε, σχετικά ε, με το τι υπάρχει ε, αν ανήκει, για να δει κανείς αν ανήκει κάπου, αν θέλει να εντυπωσιάσει ε, κάποιον. Όλοι έχουμε ε, γνωρίσει αυτό το συνέστημα του μη ανήκει, του να μην ανήκεις πουθενά. Και δεν ξέρω πώς κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει τις, τις προσμονές της κοινωνίας, πώς να ασχοληθεί κανείς με το «ον» του, το ανδρικό «ον», όταν δεν συμμορφώνεται προς την εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι για αυτόν. Ε, τι, ε, τι ε, πολιτικές κανείς χρησιμοποιεί, τι συμπεριφορές για να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, για να μην αντιφάσκει με την εικόνα που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό του. Έχουμε λοιπόν πολύ περιορισμένες συμπεριφορές ε, η μελέτη του Ινστιτούτου μας για τα στερεότυπα, τα φυγήματα, περιλαμβάνει ένα παράδειγμα ενός άντρα 30 ετών από την Ισπανία που λέει πως οι φίλοι του ε, προσπάθησαν να τον πείσουν να πάει σε έναν οίκο ανοχής. Ε, δεν πήγε για λόγους ηθικούς, αλλά λέει «Μου είχαν πει ότι αυτό το πράγμα είναι ταπεινωτικό, είναι κατάχρηση, είναι εκμετάλλευση, είναι αδικία. Δεν ήθελα να λάβω μέρος σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό ήταν σαφές για μένα. Δεν ήμουν 10 ετών, ήμουν 16-17 ετών και ήξερα ότι αυτό δεν ήταν δίκαιο. Δεν ήθελα να λάβω μέρος σε μια τέτοια επίσκεψη. Αλλά αυτό είχε συνέπειες για τους φίλους μας. Όχι πολύ σοβαρές συνέπειες, αλλά είχαν ε, σημασία. Αυτοί βεβαίως ε, θριαμβολογούσαν και υπερηφανευόντουσαν όχι δημόσια αλλά σε ιδιωτικές ε, ε, συζητήσεις και με απέκλεισαν από αυτές τις ε, συζητήσεις και συνομιλίες και με έβαλαν στο περιθώριο. Τέλος της ιστορίας. Αυτό είναι το παράδειγμα κάποιου ε, που δεν ήθελε να επιτρέψει στο περιβάλλον του να του οικοδομήσει την πραγματικότητα της αρανοπότητάς του για τον εαυτό του. Αλλά μπορεί βεβαίως και να τιμωρήθηκε έτσι διότι περιθωριοποιήθηκε. Όπως μας λέει αφέθηκε στο περιθώριο. Σε, στην άλλη ε, ε, παρουσίαση αναφέρθηκε ο όρος «ηγεμονική αρενοπότητα». Θα επανέλθω σε αυτήν την έκφραση. Ε, έχουμε αυτή την ιδέα της ηγεμονικής αρενοπότητας που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο άνδρας έτσι δεν ανήκει, έχει το την συνέστημα του μη ανήκει. Ε, είναι κάτι το καταστροφικό. Αλλά τούτων λεχθέντων ας δούμε πώς αυτή, αυτό το ατομικό επίπεδο μεταφράζεται σε σχήματα πιο γενικά Περνώντας από αυτές ε, τις ε, την εισαγωγικές παρατηρήσεις ε, στα, στις πληροφορίες που έχει το Ινστιτούτο μας. Αυτός ο δείκτης ο φετινός θα είναι ιδιαίτερος ε, διότι εστιάζεται στην, ε, στην κομβικότητα, στην διατομεακότητα που δείχνει τις πραγματικότητες, την περιπλοκότητα των διαφόρων ταυτοτήτων και αλληλεπιδράσεων ε, μέσα και βλέπουμε πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις θέσεις μας ή τις μη θέσεις μας μέσα στις τάξεις των φύλων θα περιοριστώ στις απόψεις ε, που είναι οι πιο σχετικές με την σημερινή συζήτηση, παρόλο που ο δείκτης εστιάζεται στην ανισότητα μεταξύ φύλων ως ε, την ισότητα την πιο ριζωμένη, επίσης αναγνωρίζει την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα μέσα στις κοινωνίες και μεταξύ των φύλων ε, και βεβαίως και τις διάφορες πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τους κινδύνους ε, διακρίσεων που δεν βασίζονται μόνο στην διαφορά φύλων. Γι' αυτό αρχίσαμε να εργαζόμαστε με την προσέγγιση αυτή της διατομεακότητας και θα σας δείξω ένα διάγραμμα που ίσως το γνωρίζουν πολλοί από εσά. Το προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας άνδρας που γεννήθηκε το 2015 μπορεί να περιμένει ότι θα ζήσει 77,9 χρόνια. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι βλέποντας αυτό το διάγραμμα την διαφορά, την διαφορά ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη το προσδόκιμο ζωής μπορεί να περάσει από 80,4 στη Σουηδία σε 69,2 χρόνια στην Λιθουανία. 11 χρόνια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που ζει στη Σουηδία και στη Λιθουανία. Το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο στην Εστονία, στην Λιθουανία και στην Λετονία περίπου 10 χρόνια για στην κάθε χώρα. Και εδώ βλέπουμε την ε, κόκκινη γραμμή που αναφέρεται ε, στους άνδρες και την μπλε γραμμή στο διάγραμμα που αναφέρεται στις γυναίκες. Ενώ η διαφορά στην Ιταλία και στο Λουξεμβούργο είναι μόνο 4 με 5 χρόνια, ακόμα και 3,3 χρόνια στις κάτω χώρες. Το βιολογικό επιχείρημα, δηλαδή ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, δεν εξηγεί γιατί υπάρχει η διαφορά ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη που ανέρχεται μέχρι τα 10 χρόνια. Υπάρχουν επίσης ε, και άλλα στοιχεία σημαντικά που πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ όταν ασχολούμαστε με το προσδόκιμο. Η εκπαίδευση, η παιδεία που έχει σημαντική επίπτωση στο προσδόκιμο ζωής. Στην Ευρώπη 2015 διαφέρει μέχρι 15 χρόνια σε ένα κράτος μέλος ανάμεσα στους ανθρώπους με λίγη μόρφωση και σε αυτούς που έχουν ε, ανώτερη μόρφωση, όπως και στην περίπτωση της Σλοβακίας. Μιλώντας για το προσδόκιμο ζωής αναπόφευκτα μπορεί να μιλήσουμε για την ε, συμπεριφορά ε, των ανθρώπων σε σχέση με την υγεία. Ορισμένοι τρώνε φρούτα, λαχανικά και κάνουν φυσική άσκηση, δραστηριότητες που βελτιώνουν την υγεία. Ενώ το κάπνισμα και ο τα υπερβολικά αλκοολικά ποτά είναι επικίνδυνα και υποβαθμίζουν την υγεία. Οι άνδρες είναι πιο εκτεθειμένοι σε επικίνδυνη συμπεριφορά από τις γυναίκες. Ε, το ποσοστό των ανδρών ε, που έχουν καλή φυσική δραστηριότητα ή που τρώνε αρκετά φρούτα και λαχανικά είναι ε, υψηλότερο το ποσοστό από αυτό των γυναικών, 42% για τους άνδρες, 36% για τις γυναίκες. Βλέπουμε ότι η ανώτερη εκπαίδευση και το ανώτερο εισόδημα οδηγεί τους άνδρες και τις γυναίκες σε περισσότερη ε, φυσική δραστηριότητα και ε, πέφτει με την πάροδο των ετών η φυσική δραστηριότητα. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ε, οι συμπεριφορές ε, κινδύνου όπου υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες αρκετά σημαντικές στην Ευρώπη και εδώ βλέπουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση νοπνεύματος στην Ευρώπη όπου ε, είναι αλήθεια μόνο για το εν τρίτον των ανδρών που έχουν μεσαία και ανώτερη εκπαίδευση και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Εν τρίτον ε, των ανδρών ε, πίνουν υπερβολικά. Επίσης βλέπετε εδώ στα δεξιά τον παράγοντα τον εισοδηματικό που έχει σημασία. Περνάω τώρα στο κάπνισμα, που είναι μια άλλη συμπεριφορά επικίνδυνη σε σχέση με την υγεία. Είναι πρόβλημα για πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες στην Ευρώπη, αλλά εδώ και πάλι εξαρτάται πολύ από την ομάδα αυτοί που έχουν χαμηλή μόρφωση και μέση μόρφωση ε, καπνίζουν περισσότερο από αυτούς που έχουν ανώτερη μόρφωση και αυτό ισχύει και για το εισόδημα. Όσο ψηλότερο το εισόδημα τόσο χαμηλότερο το κάπνισμα. Όπως είδαμε στις προηγούμενες εικόνες και στην προηγούμενη παρουσίαση η παιδεία είναι από τους σημαντικούς παράγοντες που προσδιορίζει την ε, τα αποτελέσματα για τις ζωές των γυναικών και των ανδρών. Και είδατε στην προηγούμενη ε, διαφάνεια πώς προσδιορίζεται η επικίνδυνη συμπεριφορά ως προς την υγεία. Σε σχέση με την εκπαίδευση βλέπουμε ότι χάνουν σιγά σιγά οι νέοι. Ε, βλέπουμε ότι διατομεακά αν δούμε το φύλλο και την ηλικία βλέπουμε ότι στις παλαιότερες γενές οι άνδρες και οι γυναίκες τώρα έχουν περισσότερη τριτογενή εκπαίδευση ενώ τώρα έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Ενώ έχουμε ε, γυναίκες 30-34 που έχουν ήδη φτάσει το στόχο της Ευρώπης 2020. Οι άνδρες με τριτογενή εκπαίδευση της ίδιας ομάδας ηλικίας έχουν 9% χαμηλότερα αποτελέσματα και αυτό διευρύνει ε, το χάσμα μεταξύ των φύλων από το 2005 όταν ε, η διαφορά ήταν 4%. Η ανώτερη εκπαίδευση είναι χαμηλότερος κίνδυνος φτώχειας ε, για τις γυναίκες. Η φτώχεια ένδια επηρεάζεται από την εκπαίδευση. Αυτό το διάγραμμα μας δείχνει ποιος επηρεάζεται και κατά πόσο επηρεάζεται ε, και μπορεί να εκτεθεί στον κίνδυνο της φτώχειας βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος φτώχειας που είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από το φύλλο είναι οι ε, άγαμοι, είναι οι μονογονικές οικοδένειες, οι ε, γυναίκες, αυτοί που έχουν ειδικέ ανάγκες όταν εξετάσουμε την κατάσταση των μονογονικών οικογενειών, των μητέρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και αυτό ισχύει ε, πολύ περισσότερο για τους άνδρες που έχουν γεννηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 38%. Και αυτό είναι σημαντικό διότι ε, οι προσμονές του να είναι κανείς ένας πάροχος φροντίδας στην ε, κοινωνία, οι προσμονές αυτές ε, είναι υψηλές, οι ελπίδες αυτές. Και οι επιλογές είναι σημαντικές. Και περνάω τώρα στο τελευταίο μέρος που έχει σχέση και με την προηγούμενη παρουσίαση, μερικά από τα αποτελέσματα από έναν ε, τομέα είδα, έδειξα ότι σε άλλους τομείς βλέπετε τις ε, διακυμάνσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες ανδρών. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι σε σχέση με τον χρόνο, τον τομέα χρόνο, παρά τις διαφορές σε άλλους τομείς, φαίνεται ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ διαφόρων ομάδων ανδρών δεν ξοδεύουν αρκετό χρόνο για την φροντίδα των αγαπημένων τους, των, ε, της γυναίκας τους, των παιδιών τους, της οικογένειάς τους. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει περαιτέρω να μελετηθεί. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και να πω ότι αυτά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες και ένας ο οποίος συμφωνεί με τα αρνητικά στερεότυπα και τα, τις ατομικές επιλογές είναι βεβαίως ότι πρέπει τα στερεότυπα αυτά να τα εξετάσουμε σε επίπεδο ε, κοινωνίας και να μην είναι η βάση των διακρίσεων. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Έρικ Μέλλαντερ, καθηγητής ε, στο τμήμα ερευνών για τις διενέξεις του Πανεπιστήμιου της Σούψαλα στη Σουηδία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε λίγο για την έρευνα που κάνουμε στην Ούψαλα. Θα ήθελα να αναφερθώ όλος ιδιαιτέρως στους άντρες και στη βία, ε, την βία των ανδρών, όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα του τι σημαίνει να είσαι άντρας. Ο τίτλος είναι ε, η, τιμή του αρσενικού, και σχετική ιδεολογία και η βία. Το σημείο αφετηρίας είναι ότι γενικότερα διαχρονικά στις διάφορες κοινωνίες έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι άντρες είναι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ασκούν βία. Είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό το στερεότυπο δηλαδή είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Ορισμένε φορές θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Και δεν κοιτάζουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και αυτό ισχύει και για την νόμιμη βία, ας πούμε, αυτή που ασκεί δηλαδή ένα στρατός ή η αστυνομία, που είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία αρσενική, αν και αλλάζουν τα πράγματα τελευταία, παραμένει όμως κατά μεγάλη πλειοψηφία ε, προνόμιο των ανδρών, και η παράνομη βία, ας πούμε, η σωματική βία σε μια σχέση, στην ενδοοικογενειακή βία, οι εγκληματίες, οι τρομοκράτες, οι εξεγερμένοι, ε, τα λοιπά. Ταυτόχρονα όμως οι περισσότεροι άνδρες δεν πολεμούν, δεν σκοτώνουν κάποιον, δεν ασκούν βία. Ακόμα και σε κοινωνίες που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από μεγάλα ποσοστά βίας, όπου υπάρχουν εμφύλιος πόλεμος, ακόμα και σε, ε, σε χώρες που βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο. Είναι, είναι μια μειοψηφία ανδρών που πολεμούν. Και βεβαίω όταν μιλάμε για τις ε, κοινωνίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βεβαίω η μεγάλη πλειοψηφία ε, όσων ε, των δραστών βίας είναι άντρε, αλλά οι περισσότεροι άντρε η μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών δεν έχει ποτέ διαπράξει πράξεις βία. Έτσι λοιπόν υπάρχει κάτι εδώ που συνδέει τους άντρες με τη βία. Κάτι που έχει να κάνει με τον, τον ανδρισμό, με τον, τον, το αρσενικό. Όμως αυτό ισχύει για κάποιους άνδρες ή ισχύει κατά προτεραιότητα για κάποιους άντρες και όχι για τους περισσότερους. Και εμείς προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό στην έρευνά μας. Πώς, εξηγεί Πώς εξηγείται αυτή η συμμετοχή των ανδρών στη βία. Οι προηγούμενες έρευνες έχουν συλλέξει πολλά στοιχεία για το πώς οι άνδρες αντιλαμβάνονται την ε, συνθήκη τους, ότι είναι άνδρες δηλαδή, ότι πώς αναλαμβάνονται τον ανδρισμό τους. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, επηρεάζει τη συμπεριφορά και επηρεάζει ιδιαίτερα την βία συμπεριφορά. Ένας άντρας λοιπόν που θεωρεί, που πιστεύει σε αυτό το αρνητικό στερεότυπο, ότι τι σημαίνει να είσαι πραγματικός άντρας. Εκεί υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι άντρες το πιστεύουν περισσότερο, κάποιοι άλλοι ταυτίζονται με άλλους τύπους ε, αρσενικότητας, όμως οι άντρες οι οποίοι περισσότερο υιοθετούν αυτήν, αυτό το στερεότυπο του, του ανδρισμού είναι και πιο πιθανό να έχουν η συμπεριφορά. Εάν του ζητήσει κανείς, το ρωτήσει κανείς αν συμφωνούν με την, το, βασανισμό ε, υπόπτων τρομοκρατίας, είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν. Επίσης, άντρες με αυτή τη συμπεριφορά αυτοί δηλαδή που ταυτίζονται με αυτού του είδους τον ανδρισμό είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν και σε εγκληματικού τύπου βία ενδοικογενειακή βία ή και βία έξω στον δρόμο βία εγκλήματα αυτοί οι τύποι ανδρισμού λοιπόν ε, συνδέονται επίσης και με την ανάληψη ρίσκου αυτοί οι άντρε συχνά είναι αυτοί που παίρνουν και τα μεγαλύτερα ρίσκα σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία πώ ταυτίζει, ταυτίζει το κάθε άντρα με τις διάφορες, τα διάφορα στερεότυπα περί ανδρισμού. Αυτό επηρεάζει και τη στάση του και τη συμπεριφορά του απέναντι στη βία γενικότερα. Έτσι λοιπόν μαζί με του συνάδελφου, τον Είναι Μπιόρνεγκουρ και τον Κορνέλιο βίνε στην Ουψάλα, έχουμε κάνει μία μελέτη που θα παρουσιάσουμε σύντομα όπου ε, επεκτείνουμε αυτή την έρευνα ε, για τη σημασία του ανδρισμού ε, και σε ό,τι αφορά την πολιτική βία. Δεν είναι μόνο θέμα στάσης, δεν είναι μόνο θέμα εγκληματικής συμπεριφοράς, βίας συμπεριφοράς, έχει να κάνει και με τη συμμετοχή στην πολιτική βία πλέον. Αυτή είναι μια μελέτη σε πολιτικούς ακτιβιστές που έχουν δραστηριοποιηθεί στην Πανκόκ, στην Ταϊλάνδη, άνδρες μεταξύ αυτών των πολιτικών ακτιβιστών εκείνοι οι οποίοι ταυτίζονται περισσότερο με αυτά τα στερεότυπα του ανδρισμού και αυτή την ιδεολογία είναι αυτοί που συμμετέχουν και περισσότερο ε, στην, σε πράξη πολιτικής βίας στην Μπαγκοκ. Τι εννοούμε όταν μιλάμε την ιδεολογία ανδρισμού. Όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο της τιμής, της ανδρικής τιμής, δεν εννοούμε την τιμή ε, με την συνηθισμένη έννοια, ότι είναι κάποιος ο οποίος ε, ε, τιμά τη χώρα του υπερασπίζοντάς την είναι κάποιος ε, ο οποίος ε, έχει ε, φιλότιμο ας πούμε όχι, εδώ μιλάμε για την ανθρωπολογική προσέγγιση είναι κάποιος ο, του οποίου το στάτους ανεβαίνει εφόσον δείχνει σκληρότητα εφόσον είναι σκληρός Και αυτό είναι η αντίθεση σχέση με τη γυναίκα η οποία στην οικογένεια είναι ε, κατά κάποιο τρόπο ευνοχισμένη. Μιλάμε λοιπόν για μια τιμή ανδρική. Αφορά τους άνδρες. Τι πρέπει να κάνει ένας άνδρας για να είναι πραγματικός άνδρας, για να, για να υπερασπίσει την τιμή του την ανδρική. Και εδώ θέλει προσοχή, διότι κάποιος μπορεί αυτό να το υιοθετήσει σε διάφορα επίπεδα, εξαρτάται από τον καθένα και δεν είναι κάτι πολιτιστικό. Δεν είναι ότι κάποιες κουλτούρες ε, αυτή την ιδεολογία και υπάρχουν εγκλήματα τιμής και αλλού δεν υπάρχουν εγκλήματα τιμής. Κάποιοι το υιοθετούν αυτό σε όλες τις κοινωνίες. Μπορεί να βρει κανείς τέτοιους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το προσμετράμε μέσω μελετών με τους πολιτικούς αυτούς ακτιβιστές, τους ρωτάμε ε, για ζητήματα ισότητας των δύο φύλων, πώς βλέπουν τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, το ρόλο της ε, ενδοκογενειακής βίας ε, κτλ. κτλ. Ε, αυτή η ιδεολογία της ανδρικής τιμής βασίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι οι αξίες ή πατριαρχικές. ότι οι άντρες είναι, υψηλό, είναι οι ισχυρότεροι από τι γυναίκε είναι ανώτεροι και έχουν και κάποια δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν την ανωτερότητα εντό τη οικογένεια. Και υπάρχει από εκεί πέρα ένα άλλο σκέλο ε, για αυτή την ανδρική τιμή που είναι η σκληρότητα. Η ανδρική σκληρότητα. Ότι ο άντρα πρέπει να είναι σκληρό, πρέπει να μην υποχωρεί για να μπορέσει να υπερασπιστεί τη φήμη του, την υπόλοιψή του. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία τα έχει κάποιο ταυτόχρονα, εκεί είναι που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος βίας. Διότι οι πατριαρχικές αξίες μαζί με ένα μοντέλο που σου λέει ότι ο μισός πληθυσμός αξίζει λιγότερο από το άλλο μισό, από τον άλλο μισό, ότι οι άντρες αξίζουν περισσότερο από τις γυναίκες, έχουν κάποια προνόμια, αυτό ε, είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και σε άλλες ομάδες από εκεί πέρα, σε μειονότητες, ε, στους ομοφιλόφιλους, ε, δηλαδή ότι η τάδε ομάδα είναι καλύτερη από τη δική μου ομάδα. Αυτή λοιπόν η σκληρότητα από εκεί πέρα η ανδρική είναι αυτή η οποία πυροδοτεί και τη βία η οποία ασκείται απέναντι σε αυτές τις άλλες ομάδες. Αυτή είναι η ιδεολογία της ανδρικής τιμής, ο συνδυασμός των δύο αυτών ε, συστατικών. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται καθολικά, όχι μόνο στην Ταϊλάνδη. Πρέπει αυτή τη μελέτη να την διευρύνουμε είναι κάτι που μας βοηθάει να εντοπίσουμε ποιος μεταξύ των ανδρών ε, ποιοι μεταξύ των ανδρών είναι αυτοί που ενδέχεται να συμμετάσχουν σε βίες ε, ε, συμπεριφορές. Με βάση τις αναλύσεις μας δεν είχε τελικά σημασία ούτε οι πολιτικές πεπιθήσεις ούτε οι ούτε η ηλικία, ούτε η εκπαίδευση. Αυτή, αυτός, αυτή η υιοθέτηση Τη ιδεολογία τη ανθρική τιμή είναι αυτή η οποία ε, καθορίζει τη συμμετοχή στη βία. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα της βίας. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε τους άνδρες να εντοπίσουν άλλες μορφές ανδρισμού, λιγότερο βίες, να υπάρχουν κάποια ε, πρότυπα, παραδείγματος χάρη. Επίσης, ε, ας δούμε και τις, ε, τους χρήστες νόμιμης βίας, τους, στρατό μας, την αστυνομία μας. Υπάρχει ένας κίνδυνος ε, εδώ υπερβολικής χρήσης βίας. Ιδιαίτερα εφόσον οι άνθρωποι αυτοί έχουν ασπαστεί την ε, ε ιδεολογία της ανδρικής τιμής. Εφόσον αυτό συμβαίνει σε, μεταξύ των σωμάτων της αστυνομίας και του στρατού, εκεί είναι πολύ πιθανό να έχουμε υπερβολική βία. Επίση, η ιδεολογία αυτή συνδέεται όπως είπα προηγουμένω με την ανάληψη ρίσκου. Οπότε εκεί μπορεί να προκύψουν ατυχήματα. Υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, το bullying, ε, άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ιδεολογία της ανδρικής τιμής και μπορούν ε, να επηρεαστούν Αυτό βεβαίω δημιουργεί μια, ένα εχθρικό περιβάλλον για τις μειονότητες και για τις γυναίκες. Και βεβαίω είναι σημαντικό θέμα για να μπορέσουμε και στις, στις στρατιωτικές δυνάμεις μας και στις αστυνομικές δυνάμεις να προσλαμβάνουμε γυναίκες και ανθρώπους που έχουν Αλλά και γενικότερα πρέπει να αυξηθεί η λαϊκή υποστήριξη ε, για την αστυνομία και το στρατό διότι αυτές ε, οι ακραίες, ε, η ακραία ιδεολογία της ανδρικής τιμής ε, δεν συνάδει με την άποψη της πλειοψηφίας της κοινής νόμης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον. Η μεγάλη πλειοψηφία όσων ασκούν βία είναι άντρες. Αλλά και γυναίκες υπάρχουν οι οποίες ασκούν βία. Έχουμε πολλά παραδείγματα ε, γυναικών στρατιωτών ε, όμως, η συμμετοχή τους στη βία συνήθως αγνοείται ή ε, την ε, ε, περιθωριοποιούμε, θεωρούμε ότι είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι περίεργο. Σε γενικές γραμμές υπάρχει αυτή η τάση υποβάθμισης, δηλαδή της γυναικείας συμμετοχής. Ακόμα και η έννοια δηλαδή ενός πολεμιστή, ενός χρήστη βίας ε, συνδέεται ακριβώς με τον ανδρισμό. Ένας πολεμιστής εν μέρη ορίζεται ως κάποιος που διαθέτει ανδρισμό. Και τα προσόντα που έχει κάποιος πολεμιστής καθορίζουν το πόσο άντρας είναι. συμμετοχή των κυριαρχών λοιπόν αποτελεί απειλή σε αυτή την παράδοση. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα στι στρατιωτικέ δυνάμει, στην αστυνομία, αλλά και μεταξύ των ανδρών, στον χώρο εργασία, στην οικογένεια και, θέλ, και μπορεί να θέλουμε να, ε, να ξεφορτωθούμε αυτή την ιδεολογία. Αλλά κάποια στοιχεία από αυτά, αυτή την ταυτότητα του πολεμιστή είναι κάποια στοιχεία τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε. Όπω η γενναιότητα, η αυτοθυσία, θέλουμε ε, να υπάρχουν τα συστατικά αυτά, τα στοιχεία αυτά στο στρατό παραδείγματο χάρη. Και εδώ θέλει προσοχή. Θέλουμε να αποσυνδέσουμε αυτές τις θετικέ αξίες και να τι διαφυλάξουμε από τον ανδρισμό γενικότερα. Θέλουμε σύγχρονα σώματα ασφαλείας, αστυνομία, στρατό, χωρίς να υπάρχει αυτή η α, ακραία ιδεολογία της ανδρικής τιμής. Τώρα Πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε αυτό. Ένα από τα βασικά ευρήματα στη μελέτη δείχνει ότι οι κοινωνίε όπου υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι και πιο ειρηνικέ. Γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν μειώνεται αυτή η ιδεολογία της ανδρικής τιμής, η γυναίκα σιγά σιγά χειραφετείται. Υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, μειώνεται η βία, μειώνεται η υποστήριξη βίαιων πολιτικών και συμπεριφορών, αυτό είναι ένα σημείο κλειδί, όχι μόνο για τη μείωση της βίας γενικότερα στις κοινωνίες μας, αλλά και για την οικοδόμηση της ειρήνης. Και εφόσον ε, οι γυναίκες και οι άντρες ορίζονται κατά, την παράθεση ένας με τον άλλον, κατά αντίθεση, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι και τα δύο φύλλα για την προσπάθεια αντιμετώπιση του ζητήματος. Ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλάντερ για την παρουσίασή του. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη για να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Ίσως οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Νιγηρίας θα ήθελαν κάτι να μας πούν. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους εκείνους που παρενέβησαν. στην Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Φίλων. Εχθές ξανακούσαμε κάποιες ε, παρεμβάσεις, παρουσιάσεις. Ε, ήμασταν μια δύο, οποία των 7 μία έφυγε. Τρεις από το Κοινοβούλιο και τέσσερις από τη Γερουσία. Σχεδόν όλες μας είμαστε μαχήτριες για τα θέματα ισότητας των φύλων. έχουμε αντιμετωπίσει οι ίδιες πάρα πολλά τέτοια θέματα, προβλήματα, κρούσματα βίας και ελεκτικής βίας αλλά κάποιος τελικά πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να αντιμετωπίσει το ζήτημα και να ορθώσει το ανάστημά του. Ίσως τα πράγματα αλλάζουν στην Ιγυρία για τα θέματα ισότητας των φύλων και ο καθηγητής στο τέλος ίσως το αποτύπωσε σωστά. Στην Αφρική οι άνδρες θεωρούν ότι είναι ανώτεροι και ότι οι γυναίκες είναι από κάτω τους. Εγώ έχω ένα δεκάχρονο γιο και ήρθε μια μέρα και το έριξε στην οικογένεια έτσι βρώμικο όπως ήταν, του είπα γιατί δεν το καθαρίζεις και μου λέει δεν είμαι εγώ κορίτσι. Και είπε γιατί να μην το καθαρίζει η αδερφή μου που είναι κορίτσι. Και είχαμε μία συζήτηση με το δεκάχρονο παιδί και αντελήφθη πώς σκέπτεται εκείνος, πώς σκέπτεται το αγοράκι αυτό ότι είναι άντρας. Και του είπα όχι, όσο μένεις μαζί μας εδώ στο σπίτι μας, θα πλένεις τα σκεύη που χρησιμοποιείς. Γιατί αύριο αν είσαι, αν στο σχολείο, τι θα κάνεις, θα περιμένεις το πλύνει κάποιος άλλος. Εγώ λοιπόν έχω εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από το σλόγγαν που είχαν εφεύρει «He for she». Δηλαδή, να ανταλλάξει κανείς την αντίληψή του, του τι σημαίνει να είσαι άντρας ή γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι, και αν θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας και για την προέλευσή μας, πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψή μας σχετικά με τους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν, τη γυναίκα μας, την αδελφή μας και τον ανδρικό σοβινισμό που διακατέχει γενικά τη χώρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι απλώς συντροφή μας, τίποτα περισσότερο. Και σιγά σιγά στο σπίτι, στο σχολείο, στην Επιτροπή Εκπαίδευσης ε, που έχουμε στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι το παν είναι η ισορροπία δεν είναι ότι κάποιος μας έφτιαξε τον ένα άνδρα και την άλλη γυναίκα Προσπαθώ λοιπόν να επανέλθω σε αυτά που είπε ο καθηγητής στην τελευταία παρουσίαση και νομίζω, ξαναλέω, το αποτύπωσε πολύ σωστά. Ιδιαίτερα στην Αφρική, στην Ήπεθρο, σε κάποια νότια τμήματα της χώρας, ε, πιστεύουν ότι ε, κάποιες γυναίκες που δεν έχουν καν αγόρι, δεν είναι καν γυναίκες. και οι γυναίκες επίσης είναι αυτές από τις οποίες περιμένουμε να αναλάβουν και τους ε, παπούδες τους ενήλικες, τους υπερήλικες με συγχωρείτε. Το μόνο επίπεδο μέτωπο στο οποίο τα πηγαίνουμε λίγο καλύτερα είναι η, η ισορροπία των ε, μισθών. αλλά και πάλι στα κοινωνικά ζητήματα, στα ζητήματα στο σπίτι, στην οικογένεια, στη θρησκεία, στα πιστεύω των πολιτών. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την αντίληψη που έχει ο κόσμος, που έχουν οι πολίτες ε, σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον 21ο αιώνα. Ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που είχαμε την τιμή να σας παρακολουθήσουμε και να τοποθετηθούμε κιόλας. Σας ευχαριστώ θερμός. Ευχαριστώ και εγώ λέει η Πρόεδρος. Δεν, ξέρει αν, δεν ξέρω αν κάποια άλλη από εσά θα ήθελε το λόγο. Ναι. Ε, ε, ευχαριστώ. Όχι, δεν έχετε ερωτήσεις, δεν έχετε σχόλια. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη ε, του πάνελ ίσως να δώσουν μερικές σύντομες απαντήσεις, μερικές παρατηρήσεις, σχόλια. Εγώ μίλη, εγώ μίλησα για ένα ε, σοβαρό πρόβλημα, την βία των ανδρών που αφορά όλες τις κοινωνίες και όλους τους πολιτισμούς. Οι δύο άλλες παρουσιάσεις μας έδωσαν ορισμένες νήξεις ε, για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ισότητα μεταξύ των φύλων και προτάσεις για μερικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, να συμμετάσχουν παραδείγματο χάρη οι άνδρες στην παροχή φροντίδας για παιδιά και άλλης φροντίδας. Σκάντερνε, ναι, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα επίσης να πω κάτι σε σχέση με τα όσα είπατε και την παρουσίασή σας όταν μιλάτε για την αντίληψη της αρενοπότητας Υπάρχει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ήρωες στην Γερμανία και στην Αυστρία, όπου κάνουν ένα είδος, ένα σχεδίο όπου ε, εργάζονται με νέους, με μουσουλμάνους για το θέμα της ε, τιμής της, ε, του μαχίστας και θα ήθελα ε, να πω κάτι σε σχέση με τα όσα είπατε. Εργαζόμαστε κυρίως τώρα σε σχέση ε, έχουμε τους μετανάστες, με τους ετούντες άσυλο, έχουμε ομάδες διαλόγου ε, με τους άνδρες για την αντίληψη της τιμής, ε, για την βία, ε, για την πρόληψη της βίας, για την αντιμετώπιση της βίας, για την προστασία κατά της βίας. Δεν θα πρέπει μόνο να να, δω, να μιλάμε για τους άντρες, αλλά να δούμε για αυτά τα διατομεακά μέτρα τι γίνεται. Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ με αυτά τα οποία λέχθηκαν και τονίζω άλλη μια φορά ότι σε όλα αυτά όταν μιλούμε για τα διάφορα αποτελέσματα θα πρέπει να δούμε πέραν των φύλων. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Να δεν υπάρχουν ερωτήματα ή σχόλια. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες ε, για αυτές τις πολύτιμες συνεισφορές ιδιαίτερα τον τομέα πολιτικής που οργάνωσε ε, αυτήν την εξαιρετικά, το εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαστήρι. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Να σας πω ότι η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα στις 16 Οκτωβρίου. Ναι. Τη Επιτροπή Γυναικών, έτσι, 16 Οκτωβρίου, το απόγευμα. Και τώρα ένα, ένα σύντομο διάλειμμα ε, έω τις 5, λέει η Πρόεδρος, συγγνώμη, συγγνώμη, διορθώνει 4 και μισή, 4 και μισή, κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Γυναικών και της Επιτροπής Ίντα. Τέσσερις και μισή.